przewodniczący! Hello. No. Yeah. No. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Τι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. The hall. Dear colleagues, let me start the sitting. Ας ξεκινήσουμε συνεδρίαση. Καθίστε στις θέσεις σας παρακαλώ συνάδελφοι. Λοιπόν, κηρύσω την συνέχιση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διακόπησαν στις 16 Δεκεμβρίου 2010. Τα πρακτικά της 16ης Δεκεμβρίου είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν σχόλια, δεν βλέπω σχόλια. Τα πρακτικά θεωρούνται λοιπόν εγκεκριμένα. Έχω κάποιες πληροφορίες να σας δώσω. Πέντε σημεία έχω να θίξω. Στις 27 Ιανουαρίου θα γιορτάσουμε την 66η επέτειο της απελευθερώσεως των συγκεντρώσεων στα Birkenau και Auschwitz, των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Και κάθε χρόνο θυμόμαστε τα θύματα αυτών των στρατοπέδων. Αυτό είναι κάτι που μας δίνει ελπίδες για το μέλλον, ότι στην Ευρώπη δεν θα ξαναδούμε τέτοιους εφιάλτες στο μέλλον. Μετά, στις 13 Ιανουαρίου, η Λιθουανία γιόρτασε την επέτειο της ε, ματηρής Κυριακής όπου ο Σοβιετικός στρατός προσπάθησε να ανατρέψει την κυβέρνηση της Λιθουανίας που είχε εκλεγεί δημοκρατικά. Είναι πλήρη μέλη τώρα του ΝΑΤΟ, η Λιθουανία, η Λιθουανία. Εκφράζουμε και αλληλεγγύη προς τη Λευκορωσία σήμερα που είναι γείτονές μας, οι Λευκορώσοι, και περιμένουν την ελευθερία και τη δημοκρατία στην πατρίδα τους. Στις 23 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση προσεχώρησε, στη, υπέγραψε την σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες. Αυτή η συνθήκη μαζί με τις αντίστοιχες στρατηγικές που έχει ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταστήσουν δυνατή την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για περίπου 18 εκατομμύρια ανθρώπους με αναπηρία που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επόμενο σημείο να σας θυμίσω ότι ανησυχούμε πάρα πολύ λόγω της εξαφανίσεως ενός Κινέζου που ήταν μέλος της αντιπολιτεύσεως βασανίζεται ε, Συζητήσαμε επανειλημμένα την υπόθεση του κυρίου Ζέγκ και καλώ την κινέζικη κυβέρνηση να αποκαλύψει πού κρατείται και ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Τέλος, μετά από την τελευταία μας σύνοδο, πριν, το, πριν τα Χριστούγεννα, έχουμε τώρα την Ουγγρική ε, Προεδρία, μετά τη Βελγική, και θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα της Ουγγρικής Προεδρίας κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου Έχουμε και σημαντικά άλλα πολιτικά γεγονότα, εκλογές στη Λευκορωσία και αυτά που να τα συζητήσουμε. Και η αναταραχή στην Ινδονησία, συγκρούς με την αστυνομία και είχαμε και φυσικές καταστροφές που συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες σε όλο τον κόσμο και θα θέλαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς, τα, προς οικογένειες των θυμάτων αυτών των θεομηνιών και προς τις κυβερνήσεις των χωρών που έχουν πληγεί από αυτές τις φυσικές καταστροφές. Έχω και άλλη πληροφορία να σας δώσω. Η ομάδα των Πρασίνων ζήτησε ο κύριος Ίντρεκ Τάραντ να ε, πάρει τη θέση του στην αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ αντικαθιστώντας τον κύριο Μπουτικόφερ. Έχετε σχόλια? Δεν βλέπω να υπάρχουν σχόλια. Οπότε έχουμε εγκρίνει αυτό τον διορισμό. Τώρα, όσον αφορά την ε, ημερήσια διάταξη, η τελική ημερήσια διάταξη υιοθετήθηκε από την διάσκεψη των Προέδρων στις 13 Ιανουαρίου. Έχει διανεμηθεί. Έχετε μπροστά σας την ημερήσια διάταξη. Προτάσεις για αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Δευτέρα. Η ομάδα των Πρασίνων Κύριε Πρόεδρε, δράτω με ευκαιρίε για την ημερήσια διάταξη να ζητήσω επίσημα η Λέδη Άστον να έρθει στην Ολομέλεια, να έρθει στο Κοινοβούλιο να μας μιλήσει για το τι έκανε και τι θα κάνει σχετικά με αυτά που συμβαίνουν.